Πρέπει να μάθετε να ακούτε και άλλες γνώμες από εκείνους που σας αρέσουν. Η περισσότερη δήλωση ήταν δήλωση απάντηση σε κάτι που λέγεται χθε. Αυτό ήταν ο κανόνα με τον οποίο εντάξει δεν ήταν διαδικαστικό. Το διαδικό σα ήταν εκτό τόπου και χρόνου. Περνάμε στην ψηφοφορία τώρα. Προβλέπει την ψηφοφορία επί τη έκθεση κυρία Βαλεάν σχετικά με την ανακοίνωση στην Επιτροπή των Επενδυτικών Σχεδίων σε Ενεργειακή Υποδομή εντό Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Προχωράμε πρώτα σε ένα μπλοκ τροπολογιών της Επιτροπής. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 327 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 41 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 59. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 77. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 74. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 78. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Τροπολογία 79. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 79. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 331 ψήφους κατά. Τροπολογία 53. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 80. Σε δύο μέρη μόνο το δεύτερο μέρος με ονομαστική κλίση. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας οφορίας. Απορρίπτεται με 348 ψήφους κατά. Τροπολογία 54. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 81. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 75. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 76 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Καταπίπτει. Πάμε τώρα στην ψήφο επί της αναθεωρημένης πρότασης. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται και τέλος με ονομαστική κλίση η ψήφος στο νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 551 ψήφους. Συγχαρητήρια στην κυρία Βαλεάν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο.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 Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία των έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με την κατάσταση στην Ουκρανία. Σας επισημαίνω ότι η πρόταση ψηφίσματος ε, Β7-115-2010 έχει αποσυρθεί. το αρχικό κείμενο της παραγράφου 4. Υπάρχει μία προφορική τροπολογία κυρίου. του κυρίου Πρέντα. Κύριε Πρέντα, έχετε το λόγο. Mulțumesc, domnule președinte. Mersi, Euh, euh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να υποβάλω την εξή ε, τροπολογιστά από τι Ουκρανικέ αρχέ που ε, δεν έχουν επικυρήσει τη Συμφωνία Πλαίσιο του Συμβουλίου τη Ευρώπη για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και των Ευρωπαϊκή Χάρτα των Μειονοτήτων να κατεβάλουν περισσότερη προσπάθεια να τίνουν χείρα προ τι μειονότητε τη χώρα ε, ζητώντας να πάρουν μέρο περισσότερο στην πολιτική εξέλιξη τη χώρα και να σεβαστεί την εκπαίδευση στη δική του γλώσσα. Ο λόγο είναι πολύ απλό. Είμαστε σε μετεκλογική περίοδο και πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι η πολιτική εξωτερική τη Ένωση στηρίζεται στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Περί αυτού πρόκειται. Ευχαριστώ. Έχει αντίθεση στην κατάθεση αυτής της προφορικής τροπολογία. Όχι, περνάμε στην ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται το αρχικό κείμενο με την προφορική τροπολογία μετά την παράγραφο 4. Μετά την παράγραφο 8, τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο της τροπολογίας 11 με συγχωρείτε. Στο 14. Ο κύριος Γκάλερ έχει μια προφορική τροπολογία. Κύριε Γκάλερ, έχετε το λόγο. Είναι για το δεύτερο κομμάτι, αλλά ε, πείτε τι τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εάν γίνει δεχτή η προφορική τροπολογία, δεν χρειαζόμαστε κατά τμήματα ψηφοφορία. Λέγεται, καλή την Επιτροπή να εφημεθεί την αναγκαίο πρόγραμμα 2011-2013 με την ε, ατζέντα της σύνδεσης. Γιατί στο κείμενο που είχαμε αρχικά είναι αντίστροφο και δεν είναι σωστά έτσι. Εάν δεν υπάρχει αντίθεση στην κατάσταση αυτής της τροπολογίας, τότε δεν προχωράμε σε split vote. Θα ψηφίσουμε όλη την παράγραφο με μία ψήφο. Επομένως, προχωράμε στην ψήφο της παραγράφου 14. Ποιοι είναι υπέρ? Ποιοι είναι κατά? Αποχές εγκρίνεται. Τώρα ο κύριος Γκάλερ έχει μια προφορική τροπολογία στην παράγραφο 15. Κύριε Γκάλερ, έχετε το λόγο. Ναι, πρόκειται για μια διόρθωση εξουσία. Γιατί όπως υπάρχει η διατύπωση αυτή τη στιγμή είναι σωστό. Στο αρχικό κείμενο δεν ήταν σωστή αναφορά. Δεν χρειάζεται να το διαβάσω. Έχετε το κείμενο μπροστά σας. Προχωράμε στη ψηφοφορία. Ε, παράγραφος 15 με την προφορική τροπολογία. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τελική ψήφος επί του ψηφίσματος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία των έξι προτάσεων ψηφίσματος σχετικά με τη 13η Σύνοδο του Συμφουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εχθών. Ο κύριος Σαλαφράγκα θέλει σε αυτό το σημείο να πάρει το λόγο. Κύριε Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χθες κατά τη συζήτηση του σχεδίου που του κειμένου πρόκειται τώρα να ψηφίσουμε είπαμε ότι ήταν 42 ετών ο κύριος Αλμπανίλ που ήταν ε, ε, φυλακισμένος, πολιτικός κρατούμενος και έκανε μια απεργία πείνας διότι ήταν ε, βάναυση και αυθαίρετη η κράτησή του και είπαμε ότι θα πρέπει να καταδικάσουμε περίφραστα αυτά τα γεγονότα. Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, ε, εκ μέρους ε, του Ευρωκοινοβουλίου να στείλετε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Θανόντος οι οποίοι πρόκειται να προβούν στην κίδευσή του και επίσης θα πρέπει να γίνει ένα διάβημα προς τις κουβανικές αρχές ο δε πρόεδρος της ε, Επιτροπής για τα ανθρώπινα δικαιώματα Λισάρδο Σάντσαθ το θεώρησε ότι είναι κάτι σαν ανθρωποκτονία ε, Θα πρέπει επομένως όσοι είναι καλόπιστοι να προβληματιστούν από αυτό το οποίο έγινε και να υιοθετήσουμε και εμείς και το Συμβούλιο κάποια εξωπρεπή θέση. Και θα πρέπει οι ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα να είναι προπόθεση των σχέσεών μας με αυτή την, ε, με αυτή την με αυτή τη χώρα, γιατί βλέπουμε ότι αυτό το πρόβλημα είναι πάγιο. Ευχαριστώ. Είναι σαφές ότι θα εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας και θα μεταφέρω το έτοιμά σας και στον ε, Πρόεδρο. Προχωράμε πρώτα στην πρόσθεση ψηφίσματος ε, της ε, ΓΚΟΕ. Ε, ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τώρα πηγαίνουμε στο κοινό ψήφισμα διάφορων πολιτικών ομάδων. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Τροπολογία 2. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ο κύριος Μπροκ έχει το λόγο. Πρόεδρε, συνάδελφοι, θα ήθελα να υποβάλω μια προφορική τροπολογία για την παράγραφο 10. Να γίνει κατά τμήματα ψηφοφορία. Ε, εκεί που λέγεται ότι θεωρεί ότι η πρόεδρο τη ιδέα αυτής στο πρωτόκολλο για συμπληρωματικά πρότυπα για τον ρατσισμό κλπ. να ξεχωριστεί να ψηφιστεί συγγνώμη ξεχωριστά γιατί κατά τη γνώμη μου δεν είναι σαφές ότι εδώ μπορούμε να ανακατεύσουμε τα διάφορα πράγματα και δεν μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα ότι η διάκριση βάσει θρησκευτικών πεπιθήσεων θα πρέπει να ε, ε, είναι ισότιμη με εκείνη των άλλων διακρίσεων. Γι' αυτό θα πρέπει να το ψηφίσουμε αυτό ξεχωριστά. Αυτό που διαφοροποιεί δηλαδή τι θρησκευτικέ διασχίσει από τι άλλε. Ο κύριο Μπροκ έχει κάνει μία πρόταση για ψηφοφορία κατά τμήματα. Αυτή η πρόταση είναι χρονικά εκτός των περιθωρίων του κανονισμού. Επομένως θα πρέπει πρώτα να ψηφίσουμε εάν δεχόμαστε να τεθεί σε ψήφο αυτή, αυτό το split. Ε, ποιοι είναι υπέρ του να υπάρξει ψηφοφορία επί του split. Όχι για το split το ίδιο, την ουσία του, αλλά για να υπάρξει ψηφοφορία επί του split. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Okay, I'll have to check this electronically. I repeat to everyone. Ηλεκτρονικός έλεγχος και επαναλαμβάνω. Δεν ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή επί της ουσίας ψηφίζουμε εάν θέλουμε ή δεν θέλουμε να έχουμε καταψήματα, τμήματα ψηφοφορίας. Λοιπόν, Electronic check. ηλεκτρονικός έλεγχος. Ποιος είναι υπέρ του να ψηφίσουμε κατά τμήματα. The vote is open. The vote is closed. Πέρασε ψηφοφορίες. It is rejected. Απορρίπτεται. Με διαφορά λίγων ψήφων. Δεν θα ψηφίσουμε λοιπόν κατά τμήματα της παράγραφο 10. Προχωρούμε στη ψηφοφορία επί της παραγράφου 17. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Electronic check on paragraph 17. Ηλεκτρονικός έλεγχος για παράγραφο 17. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 316 ψήφους. Τροπολογία 5. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 19. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 20. Ποιοι είναι υπέρ. Α, ο κύριος Μπρόκ έχει το λόγο. Πρόεδρε, και εδώ θα ήθελα κατά τμήματα ψηφοφορία, παρακαλώ. Άφησε με να μιλήσω, Μάρτιν. Η διαγραφή λίγων λέξεων στην τελευταία πρόταση. Να ψηφίσουμε κρουστό εκεί που λέει. Στη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλή η σύσταση να περιληφθούν στο διάλογο της επιστημονίας από τις δύο πλευρές και σχετικές παρατηρήσεις σε πολυμερή φόρα και το καθώς και η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ψηφιστεί ξεχωριστά και θα ήθελα να διαγραφεί δηλαδή. Για διαδικασία, ποιοι είναι υπέρ του να υπάρξει split vote σε αυτή την περίπτωση. Ποιοι είναι κατά. Αποχές Απορρίπτεται, άρα δεν θα υπάρξει split vote. Και περνάμε... You have not learned your lesson, have you? We will do this the check. Να ελέγξουμε. Αν είμαστε υπέρ ή κατά του split vote στην 20, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας απορρίπτεται με 331 ψήφους κατά. Άρα προχωρούμε τώρα στην ψήφο επί της παραγράφου 20. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 27. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ψήφος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της πρότασης ψηφίσματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων σχετικά με το πρόγραμμα δράσης του ΟΗΕ για την ισότητα των φύλων. Πεκίνο 15 χρόνια μετά. Παράγραφος 6. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος τροπολογία 2 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο Ηλεκτρονικός έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος το πρώτο μέρος της τροπολογίας 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 320 ψήφους. Δεύτερο μέρος της τροπολογίας 3. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος τροπολογίας 3. Ποιοι είναι υπέρ. Χέρια. Ποιοι είναι κατά. Εγκρίνεται, but let's check. Electronic check. Second part. έλεγχος. στο δεύτερο σημείο, τρίτη τροπολογία. Ψηφίζουμε. Πέρας. Παράγραφος 10. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, αιτιολογική σκέψη ΔΕΛΤΑ. Ποιοι είναι υπέρ. Όχι, σωρίς, με δικό μου λάθο. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Αιτιολογική σκέψη ε. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη σίγμα ταφ. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη Ζήτα, Ποιοι είναι υπέρ. Τροπολογία 4. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τελική ψήφος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται και συγχαρητήρια. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία επί της έκθεσης του κυρίου Μάνκα σχετικά με τις προβλέψεις εσόδων και δαπανών για τον διορθωτικό προϋπολογισμό 1 του 2010. Τμήμα 1 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέτω το ψήφισμα σε ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 330 ψήφους. Συγχαρητήρια στον κύριο Μάνκα. Και περνάμε στην τελευταία ψηφοφορία της ημέρας. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία επί της έκθεσης της κυρίας Ντότσιαου Πετράου Νέβες σχετικά με την πράσινη βίβλο για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλλιευτικής πολιτικής. Τροπολογία 23 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 24 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 11. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 34. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία ε, ηλεκτρονικός έλεγχος στην 34 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. εγκρίνεται με 309 ψήφους. Τροπολογία 36. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Ποιοι είναι υπέρ. Α, με ονομαστική κλίση, με συγχωρείτε. Yes, yes, yes, yes, yes. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται με 365 ψήφους κατά. Παράγραφος 12. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τσεκ, παράγραφος 12. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας Εγκρίνεται με 343 ψήφους. I just want to point out to the House that I have not been wrong. Σας τονίζω ότι ούτε μία φορά δεν έκανα λάθος σήμερα. I just We can, we can check on this. I can vote I can vote on... Αυτό μπορούμε να το επαληθεύσουμε αν θέλετε. 13 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται με 295 έναντι 291. Τροπολογία 7. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 31 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. εγκρίνεται τροπολογία 35 ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά αποχές ε, ηλεκτρονικός έλεγχος παρακαλώ για την τροπολογία 35 άρχεται ψηφοφορία Πέρα σωφορίας. Εγκρίνεται με 324 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 14. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 25. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 32 με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 33. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 37. Ποιοι είναι πέρα. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Παράγραφος 47. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 56 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 57. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 25 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 75 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 32 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 26 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 33 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της Εγκρίνεται. Επομένως η 39 καταπίπτει. Παράγραφος 86. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 40. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Παράγραφος 99 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 101. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 102 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 104. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 106. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 8. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παράγραφος 111. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 114. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Παρα, ε, τροπολογία 28. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Με ονομαστική κλίση η παράγραφος 121. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 20 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας οφορία. Εγκρίνεται. Σε τρία μέρη. Η παράγραφος 124. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 22 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Το αρχικό κείμενο της παραγράφου 135. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 30 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 9. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Έλεγχος ηλεκτρονικός στην 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 310 ψήφους. Τροπολογία 2 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη ζήτα. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ΙΒ. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ΙΙ. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη ΚΑΠΑ ΔΕΛΤΑ. Τροπολογία 10. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Does anyone want to check this? Θέλει κάποιος να ανοιχθεί αυτό αιτιολογική σκέψη ΚΘ σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Τροπολογία 5 με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Πέρας. Απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη μη έψιλον σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο μέρος ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη μη ζήτα ποιοι είναι υπέρ ποιοι είναι κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα περνάμε στην τελική ψήφο με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 356 ψήφους υπέρ, 50 κατά, 65 αποχές. Συγχαρητήρια. Okay. Make the announcements now. Yeah. Okay, well. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν προχωρήσουμε στην αιτιολόγηση ψήφου, έχω να σας κάνω μερικές ανακοινώσεις. Έχω λάβει από το Συμβούλιο τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση μαζί με το σκεπτικό που το οδήγησε στην έγκρισή τη καθώς και την θέση της Επιτροπής. Ο τίτλο θα ανακοινωθεί στα πρακτικά της παρούσα συνεδρίασης. Η προθεσμία των τριών μηνών την οποία διαθέτει το Κοινοβούλιο προκειμένου να αποφανθεί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 Προχωράμε στις αιτιολογήσεις ψήφου. Ε, πρώτα για την έκθεση Βαλεάν. Το λόγο έχει ο κύριος ε, Μπάλτσο. Κύριε Μπάλτσο, έχετε το λόγο. Ε, Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα μια, παρακαλώ, διακοπή δύο λεπτά. Δύο λεπτά διακοπή. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα έχουμε επεξηγήσει ψήφου. Όσοι είναι να φύγετε, φύγετε ήσυχα.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 Προχωράμε σε... Προχωράμε επεξηγήσεις ψήφου έκθεση κυρίας Βαλεάν. Πρώτος ο κύριος Μπάλτσο. Για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, Πρόκειται για συλλογή στοιχείων από τα κράτη-μέλη, μια προσπάθεια ταξινόμησης των στοιχείων αυτών και να είναι και προσβάσιμα για τους οικονομικούς φορείς και πολύ σωστά παρεμβαίνει στη λειτουργία της αγοράς. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ένα ψήφισμα που έρχεται σε αντίθεση με αυτό και θεωρεί ότι ο στόχος είναι σε επίπεδο ένωσης κάθε μέτρο να είναι ουδέτερο και να μην παρεμβαίνει στη λειτουργία της αγοράς η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου δεν διδάχτηκε το δίδαγμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης και ε, εξακολουθεί να διακινεί νεοφιλελεύθερα δόγματα σε μια τέτοια στρατηγική περιοχή. Είναι απαράδεκτο να σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό εγώ ψήφισα όχι. Äh, Κύριε Πρόεδρε, η λειτουργία υποδομής στην Ένωση είναι αποφασιστική προκειμένου να έχουμε ευημερία και ταυτόχρονα ασφάλεια. Ξέρουμε ότι η ενεργειακή πολιτική είναι ουσιώδης για την ασφάλεια και γι' αυτό το λόγο επιβάλλεται το Ευρωκοινοβούλιο και να συμμετέχει στη συζήτηση αυτή και να μπορεί να συμμετέχει στις αποφάσεις, να είναι πραγματικός συνομοθέτης. Γι' αυτό ζητώ από την Κομισιόν να σταματήσει την πολιτική που μπλοκάρει και να αφήσει το Κοινοβούλιο να παίξει το ρόλο του. Ε, για ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σωστή αυτή η ιδέα καθεαυτή και επομένως θα πρέπει να τονίσουμε την περιβαλλοντική πτυχή αλλά να έχουμε κάποια συνέπεια στα όσα λέμε όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος. Θα πρέπει τα επιχειρήματα τα οποία χρησιμοποιήσαμε για τον ένα πετρελαιαγωγό να τα χρησιμοποιήσουμε και τώρα. Εάν λοιπόν στηρίξουμε αυτό το έργο, να δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι στην πολιτική δεν θα πρέπει κανείς να είναι φαρισαίος και υποκριτής. Γιατί νομίζω και τέτοιο συνέβη. Eh, na začiatku v roku 2009 sa ukázalo že eh, európska únia a členské štáty si nie sú schopné vzájomne pomôcť ε, Στις αρχές του 2009 είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να βοηθήσει το ένα το άλλο όσον αφορά το φυσικό αέριο αλλά και τον ηλεκτρισμό. Γιατί είχαμε αυτά τα δύο συστήματα ε, τα οποία ήταν ασύμβατα μεταξύ τους. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την προμήθεια να είναι δυνατόν όλοι να παράσχουν τα στοιχεία που πρέπει σε σχέση με την παροχή ενεργείας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξέρει πού υπάρχουν προβλήματα, πού ε, το σύστημα μπλοκάρεται, πού υπάρχουν ε, ασυμβατότητες. Επομένως, θα πρέπει όποια χώρα έχει προβλήματα με το δίκτυο να μπορεί κάτι να κάνει. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να σταθούμε στο πλευρό της Κομισιόν και του Συμβουλίου όσον αφορά τις σχετικές πληροφορίες για το ενεργειακό δίκτυο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι αποδέχομαι το αποτελεσμα των εκλογών στην ε, Ουκρανία και με μεγάλη μου χαρά βλέπω ότι ο λαός ε, μπόρεσε να εκφραστεί ελεύθερα. Διότι διαπιστώσαμε ότι και οι αρχές αλλά και ο λαός θέλουν την δημοκρατία. Ελπίζω ότι με τις εκλογές αυτές θα έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα. Και έτσι θα υπάρξει μια γέφυρα μεταξύ Ένωσης και Ρωσίας. Άρα θα πρέπει να θεωρήσουμε ευτυχές γεγονός αυτές τις εκλογές. Επίσης θεωρούμε ότι κάτι πρέπει να γίνει με τις θεωρίες διαβατήρων πρέπει να καταργηθούν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ψήφισμα για την Ουκρανία είναι ισορροπημένο και παρουσιάζει μια αντικειμενική εικόνα της κατάστασης. Θα μπορούμε να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην Ουκρανία για να ξεπεράσει τις δυσκολίες που έχει και τον διαμερισμό της κοινωνίας για το μέλλον της χώρας. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ο κύριος Στέφαν Μπαντέρα αναφέρθηκε σε ένας ήρωας της Ουκρανίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό νομίζω, γιατί ο Στέφαν Παντέρα και οι οργανώσεις που συναναφέρονται ήταν υπεύθυνοι για εθνικούς καθαρισμούς κατά των Πολωνών. 20.000 Πολωνοί σκοτώθηκαν τότε. Ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην Ουκρανία, αλλά από την άλλη μεριά πιστεύω ότι αυτά τα ιστορικά γεγονότα πρέπει να παρουσιάζονται σωστά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 Σήμερα η Ουκρανία θέλει οικονομική και πολιτική σταθερότητα και γι' αυτό θα πρέπει να υποστηρίσουμε κάθε ε, μέτρο που θα ε, επιτρέψει την Ουκρανία να ξεπεράσει τα προβλήματά της. Θα πρέπει να αποστείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι είναι ανοιχτέ δηλαδή οι πόρτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία. Εάν θέλουμε την Ουκρανία να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα, θα πρέπει να αρχίσουμε καταργώντας το σύστημα θεωρήσεων διαβατηρίων και θα μπορέσουμε ε, να επιταχύνουμε το έργο μας. Ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είχα την τιμή να πάω στην Ουκρανία ως εκλογικός παρατηρητής και στον πρώτο και στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών πριν από λίγα χρόνια επίση οπότε θα πρέπει τώρα να θεωρήσουμε ότι η Ουκρανία είναι ένας εταίρος μας. Και θα πρέπει επίσης να εκτιμήσουμε τις προσπάθειες της χώρας αυτής δεν θα πρέπει να επιβαίνουμε στα ιστορικά της χώρας ε, πολύ όπως έγινε από πλευράς της ε, Άλντε που είπε ότι η Ουκρανία δεν στάθηκε στο ύψος των ε, περιστάσεων. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να μην ε, στεκόμαστε σε δηλώσεις, αλλά πρέπει να κρίνουμε τα πραγματικά περιστατικά. Θα πρέπει η χώρα αυτή να προσκληθεί να πλησιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης θα πρέπει να καταργηθεί ένας νόμος που υπάρχει τώρα στην χώρα το οποίο όπως είπα προηγουμένως ε, ε, συνάδελφος, ε, είναι δυνατόν να καταπιέζονται οι μειονότητες και όπως η Πολωνική. Την έκθεση, διότι την, το σχέδιο ψηφίσματος, διότι το θεωρώ ε, καταρχήν ότι προσπαθεί να, να αναμειχθεί στα εσωτερικά της Ουκρανίας, περιέχει αντιφατικές ε, αναφορές, είναι απαράδεκτο από αυτή την άποψη. Δεύτερον, γιατί θεωρώ ότι ο Ουκρανικός λαός μόνον οδύνη θα έχει από τη συμμετοχή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, το συγκεκριμένο ψήφισμα προετοιμάζει το έδαφος σε αυτή την προοπτική και βεβαίως θα υπάρχουν και ε, αναδιαρθρώσεις ε, σε αυτή τη διαδικασία όπως έχει γίνει σε τόσες άλλες χώρες. Τρίτον κύριε Πρόεδρε, και ένας από τους βασικούς λόγους που το καταψήφισα είναι η αναφορά στον Παντέρα. Πολύ καλά κάνει το ψήφισμα και αναφέρεται σε αυτό. Όμως αυτή η αίθουσα και η ευρωπαϊκή ένωση έχουν τεράστιες ευθύνες όταν έχουμε τέτοια φαινόμενα όχι μόνο στην ουκρανία την έχουμε και σε άλλες χώρες στις βαλτικές χώρες όπως ασφαλώς θα γνωρίζετε και είναι πραγματικά μεγάλες οι ευθύνες της ευρωπαϊκής ένωσης και του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για το ότι φτάσαμε να γίνεται αποκατάσταση εγκληματιών πολέμων. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ο κύριος για λεπτό. Ευχαριστώ. Η πολιτική ηγεσία στην Ουκρανία άλλαξε, αλλά ο λαός παραμένει ο ίδιο. Ζούνε σε μια χώρα που έχει ένα μεγάλο μέλλον και μεγάλο δυναμικό. Δεδομένων αυτών όλων, η Ένωση θα έπρεπε να συνεχίσει να καλλιεργεί τις σχέσεις με την Ουκρανία θα προσπαθήσει να έχει ένα πιο αποτελεσματικό διάλογο. Η Ουκρανία χρειάζεται βοήθεια από την Ένωση. Και δεν μιλάω για τους Ουκρανούς πολιτικούς, μιλάω για το λαό στην, Πολωνία, στην Ουκρανία. στην Ουκρανία. Λόγω της συνεργασίας με την Ένωση, η Ουκρανία μπορεί να έχει ένα θετικές επιδόσεις οικονομικά και πρέπει να πάρουμε πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ. Θα σας δώσω το λόγο κυρία Χάναν δύο φορές μία φορά τώρα για την Ουκρανία και κατόπιν ε, και για το ψήσιμο Βαλεάν. Οπότε έχει το λόγο τώρα για την Ουκρανία. Παρακαλώ. Thank you, Mr. President. <clears throat> Soviet communism was... Ο σοβιετικός κομμουνισμός ήταν ότι χειρότερο έχει υπάρξει απλώ ιδεολογία, γιατί οδήγησε σε φόνου τόσου πολλού, τόσου κόσμου και αυτό ήταν δυσανάλογο ε, σε σχέση με το πώ επέφερε η Ουκρανία. Και στην δεν αυτή η τραγωδία. Η Ουκρανία είναι μια λέξη που σημαίνει σύνορο, όριο και έτσι ισχύει μεταξύ των δύο μεγάλων μπλοκ της Ανατολής και της ε, Δύσης των δύο ανταγωνιστών, των δύο αντιπάλων δυνάμεων. Επομένω, θα πρέπει να δούμε πώ θα μπορέσουμε να είμαστε χρήσιμοι σε αυτή να τη βοηθήσουμε, ούτω ώστε να ανοίξει στι αγορέ μα. πρώτοι για έναν λαό που είναι μορφωμένο, ε, που έχει, έχει εξαγωγέ ανταγωνιστικέ. Οπότε, αν ανοίξουμε την, την αγκαλιά τη ε, Τη ε, Ένωση, τότε νομίζω ότι θα βελτιωθεί το βιωτικό επίπεδο αυτή τη χώρα. Από την άλλη μεριά, τι κάνουμε, τους πρόμους σε περισσότερη γραφειοκρατία ε, και του, δείχνουμε την άσχημη γραφειοκρατική πλευρά μας. Δεν θέλουν αυτό. Θέλουν απλώ μια ευκαιρία να μπορέσουν να πουλήσουν. Και τώρα κύριε Χάναν, ε, έχετε το λόγο επίση για ένα λεπτό για την έκθεση Βαλεάν, όπου εκ δεν είχατε συμπεριληφθεί στη λίστα. Παρακαλώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ανθρώπινη φύση λέει ότι όταν έχουμε κάτι απροσδόκητο προσπαθούμε να συντεριάξουμε τα, τα, τα, στην, στην νοοτροπία μας αυτά τα οποία έγιναν. Ας πούμε όταν δεν, όταν δεν ψηφίζουμε, όταν κάτι δεν, δεν συμβαίνει σε ένα δημοψήφισμα, ε, λέμε α, κάτι πήγε στραβά και αυτό γιατί δεν μας αρέσει το αποτέλεσμα. Αυτό συμβαίνει και με αυτή την χρηματοπιστωτική κρίση. Μα έχουμε την κρίση γιατί ξοδέψαμε όλα τα λεφτά, ξαντλήσαμε τους πόρους μας, δεν έχουμε άλλο πια πίστη, πίστοση και τώρα καθόμαστε και λέμε θέλουμε περισσότερο προϋπολογισμό κλπ. κλπ. Άρα έτσι δεν θεραπεύουμε την ασθένεια αλλά συνεχίζουμε τις αιτίες που την ε, προκάλεσαν. Έτσι έγινε και στον προηγούμενο αιώνα που οδηγήθηκαμε σε ύφεση και στασιμότητα οικονομική. Ερώτηση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Εθνών. πρώτα η κυρία Ανδρική Ενέ για ένα λεπτό. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ υποστήριξα το ψήφισμα αυτό και ήμουν μία από τις συντάξεις στην ε, το ψήφισμα και θα ήθελα να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Η έκθεση Goldstone έδειξε ότι οι έρευνες που γίνεται από, τις ενδιαφερό, ε, από τα ενδιαφερόμενα μέλη ποτέ σχεδόν δεν είναι αντικειμενικές ε, γιατί βλέπουμε ότι Κανένας δεν έκανε τελικά καλές και κατάλληλες έρευνες όσον αφορά τις ε, υποτιθέμενες, ε, τα υποθέμενα έγκληματα πολέμου. Επίσης, η έκθεση αυτή έχει αναθεωρηθεί πρόσφατα και έχει γίνει πιο αποδεκτή γιατί η γλώσσα που χρησιμοποιεί είναι λιγότερο πικρή. Αυτό που πρέπει να δεχτούμε είναι θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλακεί περισσότερο στη διαδικασία. Όχι μόνο κατά την έρευνα υποτιθεμένων εγκλημάτων, αλλά και προληπτικά. Ευχαριστώ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι, θα ήθελα εξ ονόματο τμήματο του ΕΛΚ και ιδίω του αδέλφου Ελμαμπρόκ να πω ότι πραγματικά ε, μας ε, πλήρωσε πολύ ότι το σώμα δεν δέχτηκε την τροπολογία να συμπεριλάβουμε και τις θρησκευτικέ και άλλες μειονότητες. Μου φαίνεται πραγματικά απαράδεκτο να εκφραζόμαστε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά να δεχόμαστε ορισμένοι που διώκονται για θρησκευτικού λόγους να θεωρούμε ότι δεν αξίζουν την προστασία μας. Το ότι δεν μπορέσαμε να το περιλάβουμε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον, γιατί θα πρέπει να προστατεύσουμε τις μειονότητες, άσχετα το τι ποιοντότητες είναι αυτές. Μόνο αν το κάνουμε αυτό θα μπορέσουμε να έχουμε το δικαίωμα να θεωρήσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παντού σε όλο τον κόσμο. Γι' αυτό εγώ καταψήφισα. Δεν μπορούμε να εξαιρέσουμε θρησκευτικέ μειονότητε. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. arvoisa puhemies aivan Ο κύριος Κάσλερ, όπως είπε, η ομάδα μας ήλπιζε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα στην ψηφοφορία. Δυστυχώς η πλειοψηφία του Κοινοβουλίου αποφάσισε να μην δώσει την ίδια προστασία στις θρησκευτικέ μειονότητες που είναι ίση σημασία. Η προστασία τους είναι ίση σημασία με προστασία άλλων μειονοτήτων. Η Ένωση θα πρέπει να δει αυτό το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Εθνών που είναι μεροληπτικό, δεν είναι καθόλου ουδέτερο. Εδώ έχουμε μόνο ένα παράδειγμα του πώς ε, χρησιμοποιήθηκε μεροληπτικά από άτομα που έχουν δική τους πολιτική ατζέντα και το πρόσφατο ψήφισμα κατά του Ισραήλ εκεί η Ένωση θα πρέπει να δει τι ακριβώς γίνεται στις εργασίες του Συμβουλίου. Κύριε Πρόεδρε, από το πέρας του ψυχρού πολέμου ένα επαναστατικό νέο δόγμα έχει επιβληθεί στα 200 κράτη των ΗΕ. Η ιδέα δηλαδή ότι οι νόμοι δεν θα πρέπει να προέρχονται από τους εθνικούς νομοθέτες που κατά κάποιο τρόπο συνδέονται με τους πληθυσμούς της χώρας αλλά πρέπει να επιβάλλονται από μια διεθνή τεχνοκρατία νομικών που είναι υπόλογη μόνο στη δική του συνείδηση. Αντιστρέφουμε 300 χρόνια δημοκρατικών εξελίξεων. Απομακρυνόμαστε από την ιδέα ότι ο λαός που ψηφίζει τον νόμο μέσω του, της κάλπης είναι υπόλογος και ξαναγυρίζουμε στην προσύγχρονη ιδέα ότι οι νομοθέτες θα πρέπει να υπόλογε μόνο στον δημιουργό τους ή στον εαυτό τους. Με τα εργαλεία αυτά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουμε τη δυνατότητα αυτές οι διεθνείς γραφειοκρατίες να πάνε πέραν των συνόρων των κρατομελών και να επιβάλλουν τη δική τους βούληση που δεν συμφωνεί με την βούληση του ντόπιου πληθυσμού. Και θα αναφέρω ένα χωρίο από το Τζαμπόρκ το στέλεχος των Ηνωμένων Εθνών είπε ότι αυτό που κάναμε είναι πραξικόπημα. Κινείται μαλακά και ήπια, παρόλα αυτά παραμένει πραξικόπημα. Περνάμε τώρα στην έκθεση Πεκίνο 15 χρόνια μετά, ο κύριος Παπα-Νικολάου. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της ισότητας των φύλων στην παρούσα φάση έρχεται αντιμέτωπο και με μία ακόμη πρόκληση η πρόοδος που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια από την ευρωπαϊκή ένωση στον τομέα της ισότητας κινδυνεύει να επιβραδυνθεί ή ακόμα και να αντιστραφεί από την τρέχουσα οικονομική ύφεση. οι αποτελεσματικές πολιτικές όμως για την ισότητα των φύλων μπορούν να αποτελέσουν μέρος της λύσης του προβλήματος για την έξοδο από αυτή την κρίση τη στήριξη της ανάκαμψης και την ενίσχυση της οικονομίας. επομένως η επένδυση σε πολιτικές που προάγουν την ισότητα γυναικών και ανδρών ανδρών και γυναικών πρέπει να αποτελούν βασική μας επιδίωξη και να στηριχθούν από όλους μας με σθένος ακόμη περισσότερο ακόμη πιο δυνατά στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στην έκθεση για το διορθωτικό προϋπολογισμό 2010. Ο κύριος ε, Βάνεκε για ένα λεπτό. Dank u voorzitter. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ντρέπεται για τον νέο προπολογισμό τον οποίο έγκριναμε διότι οι περισσότερες χώρες τώρα έχουν γονατίσει από αυτήν την τόσο σοβαρή οικονομική κρίση και χιλιάδες ε, ανθρώπων χάνουν τη δουλειά τους και εμείς εδώ ασχολούμεθα πώς θα έχουμε περισσότερα κονδύλια περισσότερα αυτοκίνητα που πληρώνουν οι φορολογούμενοι, περισσότερο προσωπικό. Αυτοί πληρώνουν την ύφη επομένω για αυτό το έξτρα προσωπικό το οποίο θέλουμε να, να, να προσλάβουμε και τελικά αυτό τι είναι, είναι κάποιες θέσεις για να έχουν κάποιο μισθό οι σοσιαλιστές που δεν ξαναεξελέγησαν. Επομένως είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό ότι καθόμαστε και βρίσκουμε διάφορα επιχειρήματα για να αντιλήσουμε ε, χρήματα από το κοινό κορβανά για αυτό το κοινό για δύο λεπτά ο κύριος Πόρτας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας αναφέρω ότι αυτός ο διορθωτικός προϋπολογισμός για αυτά τα 13 δις 13 εκατομμύρια ε, δεν είναι τόσο λογικός διότι ένα τμήμα αυτού του προπολογισμού θα πάει για να ενισχυθεί με προσωπικό το κοινοβούλιο ε, αντιπροσωπείες και επιτροπές θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνήθεια Λισαβόνας γιατί βέβαια ε, διευρύνσει αρμοδιότητε του Κοινοβουλίου, όμω έχουμε αυτά τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για κάποια κονδύλια τα οποία τα έχουν οι βουλευτέ, τα δικαιούνται οι βουλευτέ, τόσο ώστε να προσλαμβάνουν ε, του, βοηθού του. Όμω δεν θα έχουν 8, θα έχουν 16 του χρόνου. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι μια αύξηση υπερβολική. Να κάτσουμε και να λάβουμε υπόψη ότι του χρόνου προβλέπεται ε, αυτή η αύξηση 1.500 ευρώ για την αποζημίωση των βουλευτών. επομένω. Ε, από τα 16 πάμε στα 32 εκατομμύρια ευρώ. Απ' την άλλη μεριά έχουμε μια πάρα πολύ βαθιά κρίση με πολλή απεργία, ανεργία σε όλες τις ε, χώρες. Άρα είναι, είναι αφόρητο, είναι απαράδεκτο να έχουμε τέτοιες αυξήσεις για τους βουλευτές. Ενώ ταυτόχρονα ε, δεν έχουμε το, το θάρρος να περικόψουμε τις δαπάνες μας, το, τα έξοδά μας, αυτά τα οποία λαμβάνουμε εμείς αποζημίωση. πάμε για ε, μια αποζημίωση 300 ευρώ παραπάνω όταν έχουμε τα οδηπορικά, όταν ταξιδεύουμε δηλαδή. Και ένα σωρό άλλες, άλλες και επιδόματα. Όλα αυτά είναι απαράδεκτα. Όλες αυτά, όλα αυτά τα έξοδα, τα δικαιολόγητα, τα υπερβολικά, να τα περικόψουμε και να μην κάνουμε κάτι τέτοιο υπό τη σημερινή συγκυρία ε, είναι, είναι προκλητικό γιατί περνάνε τόσε δυσκολίε οι συμπολίτε μα. Δεν έχουν δώσει παράδειγμα προ αποφυγή αντί για μίμηση. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον κύριο Πόρτα και την κομμουνιστική ομάδα για το θέμα αυτό. Από την, σε όλη την Ευρώπη, από την Ιρλανδία στην Λετωνία, οι κυβερνήσει προσπαθούν να μειώσουν το κόστο για να μετώπισουν κρίση. Εμεί εδώ όμω αυξάνουμε τι δαπάνε μα σε μεγάλα ποσοστά και απόλυτα και ποσοτικά γιατί αυξάνουμε τα χρήματα που διαθέτουμε στους βουλευτές. Και η αιτιολόγηση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Λέγεται, ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε αυτά τα ε, χρήματα είναι λόγω των συμπληρωματικών ε, αρμοδιοτήτων που δημιούργησε η συνθήκη της Λισαβόνα. Εν μέρει είναι σωστό αυτό, αλλά όχι όπω το θέλανε οι συνάδελφοι. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυξάνει τη γραφειοκρατία για να εξυπηρετήσει τη γραφειοκρατία. Ο κύριος στόχος της ε, συνθήκης Λισαβόνας είναι να δώσει συμπληρωματική εργασία και έσοδα σε όλες τις δεκάδες χιλιάδες αυτών που έμεσα, η η έμεσα εξαρτώνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μόνοι που δεν ρωτήσαμε είναι η ε, εκλογείς. Και θα ήθελα να του το υποβάλουμε το θέμα για να δούμε κατά πόσο συμφωνούν να μα δώσουν συμπληρωματικά χρήματα την σήμερα ημέρα. μεταρρύθμιση κοινή στρατηγική πολιτικής. Το λόγο έχει ο κύριος ε, Ουσπάτσιτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Επικροτώ και εγώ την απόφαση για τους κοινούς κανόνες στην Αγία. η αλία όπως και τα άλλα είδη ζωής δεν μπορεί να ως δραστηριότητα δεν πρέπει να περιορίζονται σε ορισμένες περιφέρειες. Γι' αυτό είναι δύσκολο να πούμε ότι μια χώρα φροντίζει καλύτερα από τους σπόρους από ό,τι κάποια άλλη. Αν δούμε τα πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα μπορούμε να πούμε ότι ένα μεγάλο τμήμα ε, ε, ψαριών, ειδών ψαριών απειλούνται με εξαφάνιση. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κοινού κανόνες. Όχι σε επίπεδο ένωσης, σε παγκόσμιο επίπεδο. Γι' αυτό αυτό το βήμα της Ένωσης είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα καλό παράδειγμα για τις τρίτες χώρες. Ελπίζω η απόφαση αυτή, η κοινή αυτή ανάλυση να βοηθήσει τις αλληλευτικές εταιρείες και τις χώρες ασχέτως μεγέθους. Επίσης ελπίζω η απόφαση αυτή να βοηθήσει στην προστασία και ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση και αποθεμάτων με υπέρ. Διάννα Ντότζ. Κύριε Πρόεδρε, σήμερα δεν μου άρεσε καθόλου που χρειάστηκε να καταψηφίσω την έκθεση αυτή που έχει πολλές θετικές πτυχές για το μέλλον της αλληλείας μας. Παραμένει όμως γεγονός ότι για τη δική μου αλληλευτική ε, επιχειρηματική μονάδα της χώρας μου έχουμε συνεχώς άγγιση μεταχείριση από τους αλληλείς στη Βόρεια Θάλασσα με αφαίρεση διαρκώς ποσοστώσεων. Τέσσερα χρόνια κλείσιμο στην Ιρλανδική θάλασσα. Ο Ιρλανδικός τόλος από 40 αλλιευτικά πέρασε σε 6 και εξακολουθούμε να μιλάμε για υπερβάλλον δυναμικό. Τα εφαρμόζουμε λοιπόν κανόνες που ισχύουν για τη Βόρεια Θάλασσα, στην θάλασσα της Ιρλανδίας, είναι εκτός πραγματικότητας του τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Καλή η συλλογιστική, αλλά η, η Ευρώπη να επιβάλλει κάτι στην Ένωση χωρίς να εξηγεί ποιες θα είναι οι συνέπειες της νέας μεθόδου, γι' αυτό με ενθαρρύνουν μεν ορισμένες πτυχές της έκθεσης, αλλά την καταψήφισα. Ευχαριστώ. Η κυρία Αντρική για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, εγώ επιψήφισα την πράσινη βίβλο όσον αφορά την κοινή αλληλευτική πολιτική και ελπίζω ότι σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έβαλαν λιθαράκι στην προστασία του περιβάλλοντος και ε, κάναμε ένα βήμα θετικό για την αλληλευτική πολιτική. Ξέρετε ότι 27% των αλληλευτικών πόρων βρίσκονται στα πρόθυρα της εξαφάνισης Οπότε, εάν δεν περικόψουμε την, την αλία μας, αν δεν ψαρεύουμε λιγότερο, πρόκειται αυτά τα είδη να εξαφανιστούν. 86% είναι η δυνατότητα αύξησης των αλληλευτικών πόρων εάν περιοριστεί η αλληλεία. 80% όπως ξέρετε των ειδών τώρα βρίσκονται σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση και η sites πιστεύει ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η εκμετάλλευση. Άρα θα πρέπει οι μεταρρυθμίσεις να υλοποιούνται, όχι μόνο να θεσμοθετούνται. ευχαριστώ. Καταρχήν, θα ήθελα να σας πω ότι υπερψήφισα αυτό το έγγραφο. Η ομάδα μας συνέστησε πραγματικά να γίνει δεχτό το έγγραφο αυτό, αλλά το θέμα που ε, διακυβεύεται εδώ είναι γενικά η ηλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η κατάσταση των θαλασσών. Αυτό που εμένα με στεναχωρεί είναι ότι υπάρχει η υπερβολική αλλιεύση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει τώρα πια να σκεφτούμε πώς θα μπορούσουμε να προστατεύσουμε τα αποθέματα ούτως ώστε να μπορούμε να αλλιεύουμε και στο μέλλον. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τα φυσικά αποθέματα στις θάλασσες. Χρειαζόμαστε ένα πρόγραμμα που θα προστατεύει παραδείγματο χάνει τα φυσικά αποθέματα σολομού. Θα πρέπει να φροντίσουμε τα ψάρια αυτά να μπορούν να αναπαράγονται και στα ποτάμια για να μπορέσουν να μείνουν υγιεί τα αποθέματα. Για 11 χρόνια στο Κοινοβούλιο καταγγέλλω ε, τις επιπτώσεις της κοινή ελευθερικής πολιτικής ε, στην δική μας χώρα. Έχουμε 65% των πόρων που καλύπτονται ε, από την ελευθερική πολιτική, αλλά εμείς έχουμε 25% ποσοστώσεις σύμφωνα με το, το, το, το, σύστημα που υπάρχει. Επομένω, όλα αυτά είναι μόνο θεωρητικά τα οποία λέμε, διότι στην ουσία δεν υπάρχουν πια ψάρια Επομένως όλα αυτά τα οποία εμείς ε, λέμε εδώ πέρα δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα, θα έπρεπε να ανανεώνονται αυτοί οι πόροι και υπάρχουν κάποιες χώρες που θέλουν ε, να έχουν αυτοδιαχείριση Ισλανδία, Νορβηγία, Φόκλαντ εκεί έχουν αυτοδιαχείριση τα κράτη-μέλη και επομένως κάτι, κάτι κάνουν εδώ όμως έχουμε αυτή την κοινή διαχείριση όλοι μπορούν να πάνε παντού και ε, αυτό δεν είναι σωστό. Επομένως όλα όσα λέμε τώρα είναι θεωρητικά διότι τίποτα έχουν δέσει στα λιμάνια τα, τα ελληνικά, δεν υπάρχουν πια ψάρια. Ευχαριστώ πολύ. Τα πρακτικά της παρούσα συνεδρία θα υποβληθούν προ έγκριση στο σώμα κατά την έναρξη τη επόμενη συνεδριασής του. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, θα διαβάσω αμέσω τα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση στα πρόσωπα και στου φορεί στου οποίου απευθύνονται. Η συνεδρίαση λίγη. Καλή υπόλοιπη εβδομάδα, αγαπητοί συνάδελφοι.